Τη έκθεση Λίναρ για την ενσωμάτωση τη διάσταση του φίλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Uh, Θα αρχίσουμε με την εισηγήτρια. Έχετε τέσσερα λεπτά στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Ο απότερος στόχος ε, της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου είναι να επιτύχουμε ισότητα δικαιωμάτων στην κοινωνία. Χρειαζόμαστε λοιπόν συγκεκριμένες ιδέες πώς ε, με αποτελεσματικότητα μπορούμε να επιτύχουμε την ισότητα των δικαιωμάτων, ούτως ώστε να εστερνιστούν αυτές τις ιδέες οι άνθρωποι. Θα πρέπει να είναι φυσικό τμήμα της καθημερινής μας ζωής ε, αυτή η διάσταση του φύλου. Τι συνεπάγεται αυτό, σοβαρές αλλαγές στην νοοτροπία και στη συμπεριφορά ως προ, όχι μόνο προς τη μεταχείριση των γυναικών, αλλά ε, και στην αντίληψη της ποιότητας των ανθρώπων. Χρειαζόμαστε ε, επίσης την συνειδητοποίηση ε, της ε, τωρινής κατάστασης. Πολλές γυναίκες ενισχύουν την επιστημονική και στρατηγική βάση στοιχείων που χρειαζόμαστε ως απαιτούμενο βήμα για να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα όλων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν σε αυτή την έκθεση. Ήταν επικοδημητικότατη η συνεργασία τους τέλος Julia Awards, Πέτη Κάιν, Έλια Νοραβένεν. Θα ήθελα να τις ονομάσω και να σε ευχαριστήσω προσωπικά. Ως αποτέλεσμα ε, της συνεργασίας μας έχουμε ένα πολύ καλό ισόρροπο κείμενο. Όμως ε, για την ε, κοινή γνώμη παραμένει άγνωστο, άγνωστη και αμφιλεγόμενη έννοια η διάσταση του φύλου. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην προετοιμασία, την εκπόνηση, την υλοποίηση, την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών. Χρειαζόμαστε προγράμματα ότως ώστε να προωθηθεί ισότητα των ευκαιριών και των δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών ε, βλέπουμε τα απαιτούμενα βήματα για να αλλάξει ε, η τωρινή κατάσταση, να αλλάξει η νοοτροπία. Ε, τα ακόλουθα βήματα είναι απαραίτητα. Πρώτον, χρειαζόμαστε μια διαδικασία ώστε στο τομέα τη εκπόνηση πολιτικής να ενσωματώνεται πάγια η διάσταση του φύλου. Δεν θα πρέπει να εξαιρείται καμία πολιτική. Οριζόντια θα πρέπει να ενσωματώνεται η διάσταση. Αυτό είναι βασικό άξονα τη δράση μα. Δεύτερον, ω προ την εκπροσώπηση γυναικών και αντρών σε κάθε τομέα πολιτική, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό έχει μεγάλη επίπτωση ω προ το αποτέλεσμα. Δυστυχώ δεν ε, έχει έχει ε, συγκεκριμένη επίπτωση. Αυτή η δεύτερη έννοια, όχι τόσο όσο θα θέλαμε. Ε, Επίσης, ε, σταδιακά έχουμε αναπτύξει μία δομή για να ενσωματώνεται πάγια η διάσταση του φύλου. Όμως βλέπουμε κατακαιρματισμό και έλλειψη αποτελεσματικότητας. Χρειάζονται λοιπόν διορθωτικά μέτρα καθώς και ένας μηχανισμός αξιολόγησης και παροχής στοιχείων ούτως ώστε να μην μείνουμε μόνο στο γράμμα της νομοθεσίας αλλά έχουμε και αυτά αποτελέσματα. Και τέλος, για να προωθήσουμε την διάσταση του φύλου θα πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα, να δείχνουμε ακριβώς τι πρέπει πρέπει να γίνει, να μπαίνουμε στην ουσία. Ε, είναι αρχές εξαλλού αυτές που κατοχυρώνονται στη συνθήκη. Οι θεσμοί λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα για την εφαρμογή αυτών των αρχών. Και γι' αυτό μέσα στην έκθεση προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα διαθεσμικό δίκτυο όπου συμμετέχουν μεταξύ άλλων το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Εγώ πιστεύω ότι όσοι εκπονούν πολιτική εσωματώντας τη διάσταση θα πρέπει να αντιλαμβάνουν ακριβώ με ποιο τρόπο οι γυναίκες και οι άντρες μπορούν να υποφεληθούν από μεγαλύτερη ισότητα των δικαιωμάτων. Πόρο απέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις ε, δύο συνιστώσεις ε, της δράσης μας. Ελπίζουμε με την έκθεση να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και να αρχίσει μια αρχή, ε, μια, να δρομολογηθεί μια διαδικασία υλοποίηση, ώστε να επιτευχθούν όλο ένα και πιο φιλόδοξοι στόχοι. Σας ευχαριστούμε κυρία Μλίνερ. Τώρα θα αρχίσει η διαδικασία Catch the Eye. Πολλοί έχετε εγγραφεί στον κατάλογο θεωρητικά, γιατί έχουμε μόνο πέντε λεπτά. Θα επιτρέψω όμω και άλλοι να παρέμβουν, αλλά να είστε σύντομοι για να δώσουν την ευκαιρία και στου συναδέλφου να μιλήσουν. Mm. Ε, συγγνώμη, κυρία Σοϊντρόβα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μλίνα για την κατάθεση αυτής της έκθεσης. Είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει υποδειγματικό ρόλο, να δίνει το καλό παράδειγμα, δείχνοντας ποιες ευκαιρίες υπάρχουν ώστε πολιτικά να δράσουμε σε, με κάθε τρόπο από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολύ μεγάλο έργο απομένει ακόμα να γίνει και γι' αυτό πιστεύω ότι όσον αφορά την ανώτατη ιεραρχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτά τα θέματα και αιτήματα και περισσότερες γυναίκες να μπορέσουν να ενταχθούν στα υψηλά ε, ιεραρχικά αξιώματα και να δημιουργηθούν και ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τις γυναίκες για να επομιστούν αυτές τις ευθύνες. Αυτή η έκθεση είναι πάρα πολύ θετική και δίνει αυτή την διάσταση. Είμαι κατά ε, το ότι η διάσταση του φύλου θα πρέπει να επαφεθεί μόνο σε ένα επίπεδο ε, κάποιων μέτρων. Πρέπει υπερβολικά μεγάλο να δούμε εδώ ε, γραφειοκρατικό βάρος δημιουργείται και θα χάναμε από τα μάτια μας και τον πιο σημαντικό στόχο που πρέπει να επιτευχθεί που είναι η πραγματική ισότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Προσπαθώ να δώσω τη δυνατότητα περισσότεροι συνάδελφοι να μπορέσουν να, να παρέμβουν. Η κυρία Γκότη παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου. Αύριο, η 8η Μαρτίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα γυναικών. Και έτσι λοιπόν και επίσης και τα γενέθλια της ε, μητέρας μου. Και είναι πραγματικά σημαδιακή αυτή η ημέρα μια και διαφορετικές γενναίες εδώ εμπλέκονται για στη μάχη για τα δικαιώματα των γυναικών ιδιαίτερα σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αυτή την έκθεση που και εγώ ήμουν υπεύθυνη για την ε, ε, προώθησή της ε, για τον υποδειγματικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει θεσμικά η ισότητα των φύλων τα δικαιώματα των γενικών και η ισότητα βρισκόντουσαν στον πυρήνα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος ευθύς εξ ε, του ευρωπαϊκού εγχειρήματος στην Παγκόσμια ημέρα των γυναικών πρέπει να αξιολογήσουμε και να κάνουμε έναν απολογισμό και να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τις λήψεις αποφάσεων. Η ισότητα των φύλων απαιτεί να συμπεριλαμβάνουν και οι άνδρες και οι γυναίκες σε αυτή την προσπάθεια. Θα υπερψηφίσουμε αυτή την έκθεση που είναι θετική. Σας ευχαριστώ και εγώ. Είναι εδώ απαιτείται καλύτερη, ε, μεγαλύτερη εμπλοκή κοινωνικά υπέρ των γυναικών και από τις ίδιες τις γυναίκες. Έτσι μπορούμε να καταφέρουμε να έχουμε βελτιωμένες πολιτικές, κοινωνικά πολιτικές για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Πιστεύω ότι αυτό επίσης θα βοηθήσει τις γυναίκες να βελτιωθούν και να έχουν καλύτερες επιδόσεις στις επιχειρήσεις καλύτερες επιδόσεις ε, και οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ευρύτερες βάσεις ε, δεδομένων που θα βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να είναι πρωτοπόροι σε αυτή τη μάχη και να δίνεται η δυνατότητα στις γυναίκες να προαγάγουν ε, τα συμφέροντά τους. Όμως η έκθεση αυτή ακολουθεί και κάποιους, λανθασμένους προσανατολισμούς σε σχέση με τον εναρμονισμό, την, την σύγκληση τη της οικογενειακής και επιχειρησιακής ή επαγγελματικής ζωής. Ε, δεν πρέπει να ε, εμπλέκουμε τα, ε, τις προτεραιότητες μας. Η πολιτική των ολοκληρωτικών καθεστώτων πολλές φορές ανέμειξε τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια, την κυρία Μλίναρ, με την οποία συμφωνώ απόλυτα ότι η έκθεση αυτή και που ελπίζουμε ότι με μεγάλη πλειοψηφία θα υπερψηφιστεί είναι μια πολύ σημαντική έκθεση ιδιαίτερα ταιριάζει και με την Παγκόσμια ημέρα για τις γυναίκες. Δείχνουμε το πόσο μεγάλη εμβέλεια, πόσο μεγάλη σπουδαιότητα δίνεται στην ισότητα των γυναικών, όχι μόνο στην απασχόληση, αλλά και σε σχέση με το κοινοβουλευτικό έργο των Επιτροπών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Gender Impact Assessment, δηλαδή την αξιολόγηση της διάστασης, της ένταξης, της ισότητας στις πολιτικές μας, αλλά και την υλοποίηση του gender budgeting, προϋπολογισμό, δηλαδή διαμόρφωση προϋπολογισμού ε, με τα αναγκαία κονδύλια για την ισότητα των γυναικών. Σημαντικό είναι στην αυριανή ψηφοφορία από τα καλά λόγια να περάσουμε στις ε, θετικές πράξεις. Ε, το Gender Mainstreaming Network θα πρέπει και σε σχέση με τους κανόνες και κανονισμούς rules of procedures να προχωρήσουμε όπως πρέπει αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά που επετέλεσε. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα των γυναικών, μάλιστα. Αλλά δεν φτάνει με μια φορά που γιορτάζουμε αυτή την ε, ημέρα να πούμε ότι όλα γίνονται όπως πρέπει. Είναι μια σημαντική πρόοδος σίγουρα, αλλά υπάρχουν ανισότητες σε πολλούς τομείς ακόμα εις βάρος των γυναικών. Και γι' αυτό θα ήθελα να αναφέρω το θέμα των επιχειρήσεων και κυρίως όσον αφορά τα ηγετικά αξιώματα, τις ηγετικές θέσεις στις επιχειρήσεις. Πρέπει να τερματίσουμε με τα στερεότυπα που βλέπουμε να ισχύουν στην κοινωνία και στον τύπο και περισσότερες γυναίκες να επιτρέπεται να συμμετέχουν στα υψηλά αξιώματα στις λήψεις αποφάσεων. Θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικές οι επιχειρήσεις ε, και να μπορέσει να αυξηθεί έτσι και το ΑΕΠ με την σύμπραξη και συμμετοχή των γυναικών. Θα πετύχουμε την ισότητα μόνο όταν δεν θα χρειάζονται πλέον ούτε ποσοστώσεις υπέρ των γυναικών ούτε πρόσθετα μέτρα υπέρ των γυναικών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε για την επίπτωση του φύλου στις δημόσιες πολιτικές είναι ένα θέμα εξυγχρονισμού επίσης γιατί με διαφορετικό τρόπο βλέπουμε ότι έχει διαφορετικές επιπτώσεις στις δημόσιες πολιτικές. Πρέπει να αναλυφθούν μέτρα υπέρ της ισότητας για να διασφαλιστεί ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών που είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και κοινωνικό δικαίωμα. Δεν υπάρχει ουδέτερη ε, πολιτική όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνουμε. Γι' αυτό χαιρετίζω το ότι ζητείτε στο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπάρξει μια μελέτη για τις επιπτώσεις της διάστασης του φύλου. Θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα την κοινωνία. Μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερος ορθολογισμός και αποτελεσματικότητα στην χρήση των κονδυλίων, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό συμμερίζομαι απόλυτα αυτό το ψήφισμα και αυτές τις προτάσεις. Ευχαριστώ. Και ο Σουίπακ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Διαβάζοντας αυτή την έκθεση ε, εξεπλάγει και είδα κάποια παράξενα. Η εφαρμογή της διάστασης του φύλου πρέπει να συμπεριλαμβάνει την ευημερία και τον ΛΟΑΔ καθώς και όλων των ε, ταυτοτήτων και τίθεται και θέμα εκπροσωπήσεως γυναικών ανδρών και όλων των άλλων φιλετικών ταυτοτήτων. Ποιε ταυτότητε έχει υπόψη η συγκήτρια, αυτέ που υπάρχουν ή αυτέ που θα καθοριστούν και στο μέλλον. Και αναφέρει ότι οι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίζουν τα αγόρια, τα κορίτσια, τι άντρε γυναίκε, καθώ και άλλε ταυτότητε του φύλου. Αυτή δεν είναι αγόρια και κορίτσια τελικά, στο κάτω-κάτω. Και αναφέρεται η σημαντικό, το σημαντικό χαρακτήρα τη ουδέτερη γλώσσα όσον αφορά τη αίσθηση του φύλου. Και αναφέρεται ότι και η εκπαίδευση για τη μετάφραση και για την διερμηνία να χρησιμοποιούμε ουδέτερες φράσεις όσον αφορά το φύλλο. Δεν μπορεί να είστε τόσο σοβαρή τώρα. Κάποιο από εμά καταλαβαίνει ε, την ισότητα ανδρών και γυναικών και ότι είμαστε ίσοι. Σα ζητώ να υποστηρίξετε την τροπολογία 4 αύριο στην ψηφοφορία που παρουσιάζει μια εναλλακτική λύση όσον αφορά αυτή την έκθεση. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, Επίτροπε, ευχαριστώ εσάς όλες τις συναδέφους, όλες τις γυναίκες που πρέπει να τις συγχαρούμε για την αυριανή Παγκόσμια ημέρα των γυναικών. Όμως αυτή η έκθεση δεν θα συνεισφέρει να είναι μια ευτυχισμένη ημέρα. Δεν θα συνεισφέρει να μειωθεί η ανεργία εις βάρος των γυναικών και να αξιολογηθεί και να αναβαθμιστεί το, η εργασία τους ε, στο σπίτι, στην οικογένεια, ούτε θα πάψει η βία κατά των γυναικών μια υπερεπιτροπή στην οποία θα πρέπει να, υπο, ε, να εντάσσονται όλες οι αρμοδιότητες ε, των υπολείπων ε, επιτροπών. Θα δημιουργήσει επίσης περαιτέρω γραφειοκρατική επιβάρυνση, περισσότερα έγγραφα, όλο και λιγότερη διαφάνεια, όλο και λιγότερη Ευρώπη θα υπάρχει και όλο και λιγότερο θα λαμβάνονται υπόψη τα προβλήματα των γυναικών. Γι' αυτό δεν μπορώ να υπερψηφίσω αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Κυρία Βον Στόρκ. Um Μάλιστα, πρόκειται για την υλοποίηση της ιδεολογίας ε, για τα θέματα φύλου στην εσωτερική διοργάνωση του, ε, των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ζητείτε από πλευράς ε, των τμήματων να λαμβάνονται υπόψη και οι διαφορετικές επιλογές όσον αφορά τη σεξουαλική ζωή. Αυτό δεν χρειάζεται να το σχολιάσω. Πρέπει να δούμε τις επιπτώσεις που θα έχει. Έχει δύο αυτή η έκθεση. Ποια, ε, βλέπουμε ποια κονδύλια των φορολογουμένων διασπαθίζονται και ε, ε, εδώ βλέπουμε ότι τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται βλέπουμε ότι πολλές φορές χωλένουν. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. Kelly. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ, να ευχηθώ χρόνια πολλά στην κυρία Ward και η δικιά μου η μαμά έχει τότε γενέθλια αυτή η σύμπτωση. Ε, από το 1973 θα ήθελα να σας γυρίσω πίσω τότε ε, ε όταν παντρευόντουσαν οι γυναίκες δεν μπορούσαν πλέον να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Τότε επέμεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει αυτός ο κανόνας ε, και δικαίως. Λοιπόν, ε, έχει σημειωθεί η επιτυχία για την πρόθεση της ισότητας των δύο φίλων και συμφωνώ με αυτά που ακούσαμε. Ε, έγιναν εκλογές στην Ιρλανδία. Ένα τέταρτο ήταν οι γυναίκες από τους υποψήφιους για πρώτη φορά, 30% και ήταν πολύ κατά, ε, διότι έχουμε περισσότερες γυναίκες στο νέο κοινοβούλιο. Παρά την αντίσταση βλέπουμε ότι υπάρχει καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών και λειτουργούν τα μέτρα που αναλαμβάνουμε, χάρη στις ποσοστώσεις δηλαδή. Ευχαριστούμε και τώρα θα ακούσουμε την Επίτροπο ε, Γιούροβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτέ, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπλινέρ για το σχέδιο έκθεση ε, σε σχέση με την ε, ενσωμάτωση τη διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικότατο εργαλείο για να πετύχουμε την ισότητα ανάμεσα στι γυναίκε και στου άντρε. Το άρθρο 8 τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι σε όλε τι δραστηριότητε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποσκοπεί στην άρση των ανισοτήτων και στην προώθηση τη ισότητα ανάμεσα στι γυναίκε και του άντρε. Η διάσταση του φύλου, ενσωμάτωση διάσταση του φύλου δεν είναι επιλογή, δεν είναι κάτι προαιρετικό, είναι υποχρέωση. Όλα τα θεσμικά όργανα όπως και το Κοινοβούλιο έτσι και η Επιτροπή αντιμετωπίζουν πάγια αυτή την πρόκληση να ενσωματώνουν στην πράξη διάσταση του φύλου και διαρκώς να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα ε, της διάστασης αυτή. Η δυτή προσέγγιση όπως ε, αποκαλείται για τις στοχευμένες δράσεις αφενός ε, και αφετέρου για την ενσωμάτωση του, της διάστασης του φίλου σε όλες τις πάγιες πολιτικές, αυτή η διετή προσέγγιση έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Στην ε, προσφάτως ε, δημοσιοποιημένη έκθεση για το 2016 έως 2019 για την ενσωμάτωση διάσταση του φύλου αναφέρεται αυτή την προσέγγιση και βλέπουμε ότι η βασική αρχή είναι η ενσωμάτωση αυτής της διάστασης ε, του φύλου και αυτό ισχύει για όλες τις πολιτικές, για όλη την νομοθεσία, για όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πράξη γίνονται πάγια οι προσπάθειες ώστε να ενσωματώνεται αυτή η διάσταση σε όλες όλες τις πτυχές παρέμβασης και δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιολογούμε επίσης τις δράσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των γυναικών και ανδρών και επομίζομαστε τις ευθύνες για τυχόν προσαρμογή που χρειάζεται ούτως ώστε να προωθούμε την ισότητα των δύο φύλων και να μην διαιωνίζονται οι ανισότητες για να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή των δράσεων ενσωμάτωσης του φύλου, αναφέρεται η στρατηγική μας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολή έκθεσης το 2017 για την ενσωμάτωση του διάσταση του φύλου. Υπάρχει και διοργανική ομάδα εργασίας από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Τζάστα και καταναλωτών ε, που διαδραματίζει ζωτικό ρόλο για να ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πτυχέ τη δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, χρόνια πολλά κυρία Βόρντ, επίση και ε, καλή ημέρα των γυναικών σε όλες μας και όλους μας ε, για αύριο. Ευχαριστώ για τη συνεργασία. Ευχαριστούμε την Επίτροπο. Θα ήθελα